Ok. Je vous propose si, de commencer, si vous voulez bien. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Σας προτείνω να ξεκινήσουμε. Βλέπω να υπάρχουν πολλοί στην αίθουσα. Θα έλεγα να κοιτάξουμε να είμαστε αποτελεσματική και διεκπαιρεωτική, οπότε αν θέλετε ησύχω. Εκτός από αυτούς τους οποίους θα δώσω το λόγο στο επίπεδο της διερμηνίας σήμερα, Έχουμε γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ολλανδικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ουγγρικά και πολωνικά και ελληνικά για το πρόγραμμα εργασίας των τεσσάρων εργασιών που ασχολούνται με τα θέματα απασχόλησης. Αυτά εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Απασχόλησης, ΣΕΝΤΕΦΟΠ, Eurofon, ETF και ότσα, όσα, ε, τα οποία δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο της ε, Επιτροπής μας, οπότε μπορείτε να δείτε τη σχετική ενημέρωση και με mail. Στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να κοιτάξουμε το σημείο για τις διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Αρχή της Εργασίας. Εάν θες να μας ενημερώσεις εσύ. Βεβαίως, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ σύντομα για τις διαπραγματεύσεις για την ΕΛΑ. Είχαμε τριμερή διάλογο την Τρίτη το απόγευμα. Πολύ καλά πήγε. Προοδεύσαμε. Υπάρχουν κάποια ισονοσημασία ζητήματα σε κρεμότητα που θα πρέπει να τα σκεφτούμε σε επίπεδο Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, αλλά τα υπόλοιπα μοιάζουν ε, μια χαρά. Έχουμε επόμενο τριμερή διάλογο την Τρίτη στο Στρασβούργο και είμαστε, ε, έχουμε πολύ αυτοπεποίθηση ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την έξεταση του θέματος. Μάλλον εγκαίρος και για να σεβαστούμε, να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και από την πλευρά τη δική μας και του Ρουμανικής Προεδρίας βεβαίως και της Επιτρόπου Τάισεν. Ε, η πρόταση είχε δημοσιευτεί μόλις πέρσι το Μάρτιο. Θα είναι μεγάλο επίτευγμα να ολοκληρώσουμε, αλλά ε, κοιτάζουμε ακόμα κάποια, κάποια θέματα που είναι σε εκκρεμότητα. Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε στην Τρίτη. Ωραία λοιπόν, ωραίες ειδήσει. Δεύτερο θέμα, ο τριμερής διάλογος για το τρίτο πακέτο που αφορά την προστασία των εργαζομένων για, τις, για τους μεταλλαξιογόνους και καρκινογόνους παράγοντες. Προχώρησε ο τριμερής διάλογο με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα μπω τώρα στι λεπτομέρειε, γιατί είναι ένα θέμα αρκετά τεχνικό ω προ τις διάφορες ουσίες που καλύπτει. Έχουμε λοιπόν μια συμβαστική πρόταση αρκετά ικανοποιητική σε σχέση με την πρόταση του Κοινοβουλίου για το κάδμιο με μεταβατική περίοδο αρκετά ε, μακρά, 8 ετών. Έχουμε διαφορετικές τιμές που επιτρέπουν να σεβαστούμε τα όρια των βιολογικών τιμών που συνιστώνται. Και για τη φορμαλδεΐδη Έχουμε πάλι μεταβατική περίοδο 5 ετών, μεγαλύτερο διάστημα για τον τομέα της υγείας και της, των τελετών, των κηδιών, ώστε να μπορεί και στην περίπτωση της ε, ταφής του νεκρού και της και στις τοξικές ουσίες που μπορεί να υπάρχουν τη στιγμή της ε, ετοιμασίας του για την ταφή, να μπορεί να καλυφθεί και αυτή η ουσία. Αυτά για την οδηγία των καρκινογόνων και αλλαξιογόνων. Και θα προχωρήσουμε σε μία ακόμα συζήτηση που θα μας επιτρέψει να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες για να αποσαφινιστεί η διατύπωση. Ο κύριος Κάζα δεν είναι εδώ. Έγινε και ο τριμερής διάλογος για την εξισορρόπηση ιδιωτικού επαγγελματικού βίου. Έκτος γύρος και τελευταίος επί του θέματος συνοψίζοντας συμφώνησαν δύο μήνες γονική άδεια με αμοιβή ε, που δεν μεταφέρεται και δύο εβδομάδες με ε, άδεια ταινία που μπορεί να συνδυαστεί με την άδεια μητρότητα εφόσον το επιτρέψουν τα κράτη-μέλη. Αλλά εκεί δεν βρέθηκε ακόμα πολιτική συμφωνία. Επίση, τριμερή διάλογο για τι συνθήκε εργασία που θα πρέπει να είναι διαφανεί και προβλέψιμε. Ο κύριο ε, Καλβέ Σαμπόν είναι εδώ, οπότε σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είναι θαύμα που είμαι εδώ. και νομίζω ότι μπορώ να φέρω καλές ειδήσει στην ομάδα και στους βουλευτέ. Στις 3.30 το πρωί καταλήξαμε σε συμφωνία επιτέλου, μια συμφωνία που φαινόταν απίθανη. Επτά οδηγίες, φοβερά περίπλοκες, από πολιτική σκοπιά κυρίω, όπου η ενισχυμένη πλειοψηφία του Συμβουλίου ήταν δύσκολο να επιτευχθεί Είχαμε μια από τις μεγάλες χώρες που ήταν κατά, αλλά πίστηκε. Και από την πλευρά του Κοινοβουλίου χρειάστηκε να γίνει μεγάλη υποχώρηση. Και ασχοληθήκαμε με το νόμο πλαίσιο για τα δικαιώματα των εργαζομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίω μια οδηγία του 1991 για το right of statement τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν ήταν προσαρμοσμένο στις σύγχρονες συνθήκες και ιδίω για τα νέα είδη εργασία που χρειάζονται ευελιξία, αλλά που δεν πρέπει και να γίνονται αντικείμενο κατάχρηση. Οπότε το περιεχόμενο είναι πολύ περιπλοκό, υπάρχουν πολλά κεφάλαια, διαφορετικά σημεία με το, την υποχρέωση ενημέρωση, την ενίσχυση, την παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που πρέπει και αυτή να είναι καλύτερη νομίζω ότι μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας εξ και προ όφελο των πολιτών. Δεν θα πω των εργαζομένων, θα πω των Ευρωπαίων πολιτών για το μέλλον. Σας ευχαριστώ όλους, ε, όλη τη βοήθεια που δέχτηκα από τους βουλευτές ε, και τους συνεργάτες μας, τη γραμματεία μας ε, και τους δικούς μου συνεργάτες, τη θεωρώ πολύτιμη και ακόμα και για τους συνομιλητέ μου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου έχω να εκφράσω ευχαριστίες. Εδώ βρισκόμαστε. Τώρα οι εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών θα έχουν την ευκαιρία να το μελετήσουν και θα δουν και οι βουλευτέ κατά πόσο είναι καλό για το μέλλον των εργαζομένων. Πρόεδρο, ευχαριστώ για την ενημέρωση και ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ Πραγματικά, με τέτοια νύχτα που πέρασες, δεν πρόλαβες να κοιμηθείς φαντάζομαι ιδιαίτερα. Mm. Ε, να λοιπόν και κάποιες εκβάσεις τερμερών διαλόγων που είναι ευχάριστες από τον της Επιτροπής μας. Νομίζω ότι καταφέρνουμε να πλησιάσουμε πολύ το στόχο μας, να ολοκληρώσουμε την εξέταση των ε, νομοθετικών θεμάτων που έχουμε μπροστά μας και να μην μα προλάβει το τέλος της θητείας. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Μεταφορές και τα σχετικά ντοσιέ. Υποβλήθηκαν συμβαστικέ προτάσει από του εισηγητέ τη Επιτροπή Τραν για τα τρία σημεία του πακέτου κινητικότητα. Αναπέμφθηκαν στην από την Ολομέλεια στην Επιτροπή Τραν για να τα επανεξετάσει. Μιλάμε για την απόσπαση των εργαζομένων στον τομέα αυτό και το χρόνο ανάπαυσης αναφέρθηκαν οι κανονισμοί 1701, 1070 και 1071. Θα υποβάλουμε τα αποτελέσματα της Επιτροπή Τραν στην Ολομέλεια για την έκθεση Βαντενκάμπ, Όμως δεν έχει βρεθεί καμία συμβαστική λύση. Αφού έγινε εσωτερική συζήτηση σε όλες τις πολιτικές ομάδες και στην Επιτροπή Τραν, τώρα θα ακολουθήσουμε τη σύσταση της Διάσκεψης των Προέδρων. Τα τρία ντοσιέ θα προβλεφθούν στην ημερήσια διάταξη τη Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα για να έχουμε τροπολογίες από την Επιτροπή και οι τροπολογίε τη Επιτροπή πρέπει να υποβληθούν εγκαίρω στις 13 Φεβρουαρίου μάλλον θα περάσει το θέμα στην Ολομέλεια, οπότε για τα δύο πακέτα κινητικότητας που βάσει του άρθρου 54 έκθεση μπακ για το χρόνο οδήγηση και τη κυρία Γιαμέροβα για τους οδηγούς, τους αποσπασμένους οδηγούς, εκεί μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίε βάσει του άρθρου 54 Και γι' αυτό θα ψηφίσουμε σήμερα τι τροπολογίε τη Επιτροπή μα σχετικά. Σα προτείνω να περάσουμε απευθεία τι ψηφοφορίε των δύο αυτών σημείων. Ψηφίζουμε απευθεία ηλεκτρονικώ, διότι δύο ψηφοφορίε είναι όλε και όλε. Θα ήταν λίγο ανόητο να χάσουμε χρόνο και να μην ξέρουμε επακριβώ τι ψήφισε ο καθένα. Πρώτη ψηφοφορία. Έκθεση Τζαμπάγιοβα.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 Δεύτερη ψηφοφορία σήμερα. Μπακ. Θα ψηφίσουμε για την Ολομέλεια, εν της Ολομέλειας. Έχετε τον κατάλογο μπροστά σας, δεν θα αναφέρω όλα τα νούμερα. Α, καλά. Ένα, Αυτές είναι οι τροπολογίες. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται 30 προς 17 και μία αποχή. Σας ευχαριστώ. Et là, je vais laisser quelques minutes pour θα διακόψω για λίγα λεπτά για να μπορέσουν να φύγουν ε, ε, όσοι χρειάζεται να φύγουν και θα αντικατασταθώ από τον αρμόδιο στο Προεδρείο. So, liebe Kollegen, ich äh, denke, wir fahren fort in unserer Tagesordnung. Wir haben, es bleibt uns noch ein Punkt übrig. Und, ähm Συνάδελφοι, να προχωρήσουμε. Έχουμε ένα τελευταίο σημείο με δύο συνεισηγήτριες. Ε, την κυρία Χάρκιν δεν τη βλέπω, αλλά θα δώσω το λόγο στον Ζήκε για να μας κάνει την εισαγωγή στο θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας διαβάσω κάποιες ε, σημειώσεις που μου έδωσε η Μαριάν για, αυτό το σημαντικό θέμα στο οποίο είναι συνεισηγήτρια με τον κύριο Λάμπερτ την κυρία Λάμπερτ. That the two borders <laughs> absolutely affected by this very important issue that is. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, ακριβώς γιατί δίνει την ε, προοπτική της Επιτροπής Απασχόλησης ε, εν ώψη του Brexit. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει τελικά, αν θα είναι μισό Brexit, αν θα είναι κανονικό Brexit ή όχι. Σας τα διαβάζω λοιπόν. Καταρχάς να σας ζητήσω συγγνώμη για την απουσία μου, για προσωπικούς λόγους. Τις τελευταίες μέρες εγώ και η Τζιν Λάμπερντ και η σύμβουλοι μας έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις, έχουμε καταλήξει κάποιες συμφωνίες για μια κοινή προσέγγιση και θα σας τα διαβάσει αυτά η Τζιν σήμερα το πρωί. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και να θέσω κάποια ερωτήματα στην Επιτροπή προσωπικά πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι κρίσιμη σημασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να υπερβεί αυτά τα όρια της η πρόταση. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρά το γεγονός ότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τον Brexit και ότι εξακολουθώ να, πιστεύω, να ελπίζω ότι δεν θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση χωρίς συμφωνία. Παρόλα αυτά, έχουμε καθήκον να βάλουμε ένα δίχτυ ασφαλείας, να θεσπίσουμε ένα τέτοιο δίχτυ ασφαλείας για να προστατεύσουμε τους πολίτες που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία. Ωστόσο, αυτό το δίχτυ ασφαλείας πρέπει να είναι αποτελεσματικό και να προστατεύσει εκείνους που θα πληγούν σε περίπτωση σκληρού Brexit. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη έχουν σημαντικό ε, ε, ρόλο να διαδραματίσουν και δεν εναπόκειται μόνο στην Κομισιόν να υποβάλει προτάσεις για όλα τα ενδεχόμενα. Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για κάποιες ε, μεταβατικές περιόδους, μια περίοδο εφαρμογής, όπως θέλετε πείτε την, ώστε Ευρωπαίοι πολίτες να μην γίνουν ε, παράπλευρες απώλειες, να μην ε, γίνουν παράπλευρη απώλεια μιας κατάστασης κατά την οποία θα γίνει Brexit χωρί συμφωνία. Πρέπει να αναλυφθούν αντίστοιχε κινήσει και από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε κάθε περίπτωση το επίκεντρο κάθε νομοθεσία από την Κομισιόν και που θα συναποφασιστεί εδώ, από εμά και το Συμβούλιο, θα πρέπει να είναι ο πολίτη. Αλλά όπως είπα, Τζιν θα σας δώσει τις λεπτομέρειες σε σχέση με αυτά, οπότε δεν θα σας κουράσω εγώ με περισσότερα επιχειρήματα. Αλλά πριν σας θέσω τα τρία ερωτήματα που θέλω, πρέπει να πω ότι η ομάδα του Άλντε και ε, ο συντονιστής που είμαι εγώ, ε, συμφωνούμε απόλυτα με τα όσα σας διάβασα. Τα τρία ερωτήματα για την Κομισιόν είναι τα εξής μπορεί η Κομισιόν να αποσαμφινίσει αν θα ήταν δυνατόν να προβλεφθεί οποιαδήποτε παράταση του ε, καθεστώτος ε, ε383. Υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιες καποιες ακόμα και με την Τουρκία Υπάρχει και το άρθρο 352, το οποίο προβλέπει ακριβώ τέτοιε καταστάσει. Μια κατάσταση δηλαδή στην οποία έκτακτη ανάγκη, στην οποία απαιτείται ε, νοσιακή δράση. Επίση, η Κομισιόν μπορεί να προσδιορίσει ποιε ε, περαιτέρω δράσει θα πρέπει να αναλυφθούν από τα επιμέρου κράτη-μέλη, τα οποία θα μετριάσουν τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι πολίτε και αν υπάρχει ρόλο για ε, την ε, Κομισιόν ή για το Κοινοβούλιο στη δικασία αυτή. Θέλω να πω, να αναφερθώ δηλαδή σε ζητήματα όπως ε, επιδόματα παιδιού, επιδόματα ασθενείας κτλ. Τελευταίο ερώτημα. Η Κομισιόν έχει αξιολογήσει τον αντίκτυπο της μη εφαρμογής των κανόνων της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της Μαρία Äh, äh, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαμπόν. Να δώσω το λόγο στην Τζιν Λαμπέρτ που είναι η συνεισηγήτρια στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Μαριάν, θέλω να ευχαριστήσουμε τι άλλε πολιτικέ ομάδε για τη δυνατότητα που μα δώσαν να ε, συνεργαστούμε στο φάκελο αυτό. Όσον αφορά την ουσία τη πρόταση που συζητούμε, Υπάρχουν κάποια μέτρα έκτακτη ανάγκη σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ηνωμένου Βασιλείου εν ώψη τη 29η Μαρτίου 2019, που είναι η ημερομηνία από την οποία και έπειτα το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση λοιπόν προσπαθεί να μετριάσει κάποιε από τι ερευνητικέ επιπτώσει που θα είχε κάτι τέτοιο στου πολίτε που έχουν ε, ασκήσει το δικαίωμα που τους παρέχει η συνθήκη στην ελεύθερη κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία αυτή και αφορά τη διατήρηση ορισμένων δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης τα οποία ε, καλύπτουν αυτή τη στιγμή ε, τους πολίτες στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης βάσει του κανονισμού 883 στην απασχόλησή του, στη διαμονή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάποια στιγμή στο παρελθόν. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για αυτούς που αυτή τη στιγμή τα 3 εκατομμύρια Ευρωπαίου πολίτε που αυτή τη στιγμή ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όλου του Ευρωπαίου πολίτε που ενδεχομένω έχουν ασκήσει τα δικαιώματά του στο παρελθόν ε, σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση και την ε, κοινωνική, στην κοινωνική ασφάλεια. Ή και το αντίστροφο βεβαίω για ε, Βρετανούς πολίτες που έχουν ασκήσει τα αντίστοιχα δικαιώματα σε, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τις 29 Μαρτίου 2019. Στόχος μας είναι λοιπόν να μην υπάρξει παραβίαση αναδρομική αυτών των δικαιωμάτων. Ω συνεισηγήτριε, θα υποβάλουμε μικρό αριθμό ε, τροπολογιών τις οποίες και έχουμε αποστείλει ήδη την προηγούμενη εβδομάδα στους συντονιστές που καλύπτουν ορισμένα θέματα που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γίνει ό,τι πρέπει προκειμένου οι πολίτες να έχουν έγκαιρη και ακριβή ενημέρωση και να διατεθούν οι σχετικοί πόροι. Επίσης, ζητούμε από την Κομισιόν να συντάξει μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτής της πρότασης σε περίπτωση που χρειαστεί και να προσδιορίσει τομεί ανησυχία που έχουν αναδειχθεί και επίσης θέλουμε η πρόταση αυτή να ισχύσει με την επιφύλαξη άλλων νομοθετημάτων που θα υποβληθούν βάσει των αναγκών είτε έχουν υποβληθεί αυτή τη στιγμή οι προτάσεις αυτές είτε όχι ακόμη. Ακούσατε και στην παρέμβαση εκ μέρους της κυρίας Χάρκινγκ ότι μας ανησυχούν οι τομείς και θέλουμε να μάθουμε την άποψη της Κομισιόν για το τι θα γίνει με εκείνους που για παράδειγμα υπόκεινται σε ιατρική περίθαλψη αυτή τη στιγμή και που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 29 Μαρτίου Ποιε θα είναι οι επιπτώσεις στα επιδόματα, στην υγειονομική περίθαλψη. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης θα συνε... Ε, ε, ε, πάβει να ισχύει στις 30 Μαρτίου του 2019. Μέχρι τις 29 μπορείτε να πάτε και στον οδοντίατρο. Αλλά τι θα γίνει από τις 30 και μετά και ποιο πεδίο εφαρμογή πιστεύει η Κομισιόν ότι θα μπορούσε να υπάρξει προκειμένου να συνεχίζουν τα δικαιώματα των πολιτών να προστατεύονται, των οποίων η καθημερινότητα δεν αλλάζει βεβαίω από τι 29 Μαρτίου στι 30 θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, θα συνεχίζουν να εργάζονται. Αυτά τα δικαιώματα θα, θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μπορούν να μετακομίσουν ή να επιστρέψουν. Και επίσης, αυτό που είπε και η Μαριάν, αν δεν υπάρξει μεταβατική περίοδο, αν, περίοδος, αν δεν υπάρξει συμφωνία και αν αυτή η νομοθεσία καταστεί περιττή μετά τι 29 Μαρτίου, τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν για, κάποιο, για πολύ για κάποιους πολίτες, γιατί κάποιοι έχουν ε, εξαγάγει δικαιώματά τους συγκεκριμένα σε άλλε χώρε. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι υπήρξε κάποιος, ε, ότι υπήρξε πολίτης, ο, οποίος ε, παίρνει επίδομα αναπηρία και στην, Βρετανία και του είπαν ότι αυτό θα κοπεί στις 30 Μαρτίου. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για τους πολίτες που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Θα μπορούσαν να υποβληθούν ή να θεσπιστούν περαιτέρω νομοθετικές πράξεις. Εναπόκειται αποκλειστικά στα κράτη-μέλη και σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη-μέλη να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι περιστάσεις. Να πω και κάτι επί της διαδικασίας κύριε Πρόεδρε γιατί ε, προβλεπόταν αυτό, αυτή η συζήτηση να γίνει υπό το άρθρο 50, μια ταχεία διαδικασία δηλαδή για ε, μη αμφιλεγόμενους, μη ε, ακανθώδεις ας πούμε φακέλους, αλλά το Συμβούλιο ε, σημείωσε ότι τελικά θα, θέλει, θα θελήσει μάλλον να υποβάλει ουσιώδεις τροπολογίες, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Άρα μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την ταχεία διαδικασία προκειμένου να μπορούμε να έχουμε περισσότερη ταχύτητα και ευελιξία με τους συντονιστές γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όλη, αυτή η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί στις 29 Μαρτία ώστε να δοθεί τουλάχιστον εν μέρη μια κάποια βεβαιότητα στους πολίτες για το τι θα τους συμβεί. Γι' αυτό ε, ζητώ να εργαστούμε όλοι γρήγορα, ταχύτατα ε, και με πολύ στενές ε, χρονικές προθεσμίες προκειμένου να τα καταφέρουμε να τελειώσουμε την διαδικασία αυτή. Ωραία. Να ευχαριστήσω τις δύο συνεισηγήτριε. Να περάσουμε στους σκιώδει. Ο κύριο Σβέν για το ΕΛΚ. Ähm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τις συνεισηγήτριες για τις τοποθετήσεις τους Ακούστηκαν πολλά σωστά πράγματα. Προφανώς έχουμε τεράστια χρονική πίεση, είμαστε ήδη στο Φεβρουάριο και έχουμε χρόνο μέχρι τέλη Μαρτίου. Δεύτερο, αυτό που μου κάνει εντύπωση, κοίταξα και τι κάνουν οι άλλες επιτροπές με αυτή την κατάσταση. Σε όλες τις άλλες επιτροπές λοιπόν ακολουθεί τη ταχεία διαδικασία. Εδώ ακούω ότι τελικά μάλλον μια κάπως διαφορετική διαδικασία θα ακολουθεί. Τέλο πάντων δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εγώ πάντως για το ΕΛΚ ισχύει ότι το θέμα αυτό δεν είναι μικροπολιτικό. Πρέπει γρήγορα να βρεθούν λύσεις ακόμα, που θα καλύπτουν ακόμα και την περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία. Και η συνάδελφος Λάμπερτ ανέφερε κάποια σημαντικά θέματα τα οποία πράγματι πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εμείς ως ΕΛΚ Έχουμε συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με επικοδομητικό τρόπο, στο μέτρο του δυνατού. Και θέλω να παρακαλέσω όλους να μην, ξεχνα... να μην ξεχάσουμε ότι ο χρόνος πιέζει, πρέπει να φτάσουμε σε λύσεις. Γι' αυτό και εκφράζω κάπως την έκπληξή μου για το γεγονός ότι σε αντίθεση με τις άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ακολουθούμε εδώ την ταχεία διαδικασία, αλλά μια κάπως πιο καθυστερημένη, αργοπορημένη διαδικασία. Αλλά τέλος πάντων ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές δεν βλέπω τον ε, συνάδελφο. Α, θα έρθει. Οκ. Okay. Περνάμε στους ε, ECR. Helga Στίβενς Oké, okay, dank u wel, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές, τις εισηγήτριες για τις εξηγήσει τους. Παρόλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Βεβαίως ο χρόνος μας πιέζει και είναι πολύ σημαντικό να βρούμε μια λύση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών. Είτε πρόκειται για Βρετανοί πολίτες, είτε πρόκειται για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Ελπίζω να μην προκύψει η κατάσταση no deal ή τουλάχιστον αν κάτι τέτοιο προκύψει να προετοιμάσουμε μια εναλλακτική, τουλάχιστον να υπάρχει προστασία όσον αφορά την περίθαλψη για τους Βρετανούς και τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα και την κοινωνική ασφάλιστη θα προστατεύονται. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω ότι υπάρχει μια επικοδομητική συνεργασία από όλου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Για την ΚΟΑ βλέπω την Λίνμπαλ, όχι ούτε από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες, η ΕΝΕΦ, η ΕΡΤΕΝΤΕ. Ο κύριος Μπάλας δεν είναι εδώ ακόμα. Να δώσω το λόγο στο Γενικό Διευθυντή της Επιτροπής την απασχόληση. Α, βλέπω κάποιον που ζητάει το λόγο. Η Ντανούτα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ προσωπικά λυπάμαι πάρα πολύ που τελικά όλες αυτές οι αρνητικές συνέπειες που φοβόμασταν φαίνεται να πραγματοποιούνται. Κανείς δεν ήθελε να φτάσουμε εκεί. Πρέπει λοιπόν να βρούμε την ε, λιγότερο επώδυνη λύση. Ουσιαστικά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με όλους αυτούς τους Βρετανούς οι οποίοι εργάζονται στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα γίνει με τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Αν μπορούν να μεταφέρουν αυτά τα δικαιώματα στη Μεγάλη Βρετανία. Τι ακριβώς θα γίνει. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία δεν συντονίζονται μέχρι τώρα. Εάν υπάρξει λοιπόν σκληρό Brexit, δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν οι πολίτες επειδή ακριβώς αποφάσισαν να εργαστούν και να ζήσουν σε μια άλλη χώρα. Χρειαζόμαστε λοιπόν σε κάθε περίπτωση να υπάρξει συντονισμός και συνυπολογισμός εδώ των δικαιωμάτων. Και σίγουρα πριν το τέλος Μαρτίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα αυτά που αφορούν τουλάχιστον την περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση. Και θα πρέπει να δούμε επίσης και τις ε, οικονομικές ε, πτυχές, παραδείγματος χάρη που αφορούν τα επιδόματα ανεργίας και όλα τα άλλα επιδόματα για κάποιον παραδείγματος χάρη που επιστρέφει στη χώρα του μετά το Brexit Ξέρουμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσουν να υπάρχουν πολλοί αποσπασμένοι εργαζόμενοι. Ποια είναι η πρόβλεψη που έχουμε κάνει για τα δικά τους δικαιώματα. Η δική μας προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή προστασία των πολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Βλέπω ότι ο Γκυγιόν και θα του δώσω αμέσως το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ζητώ συγγνώμη, δεν ήμουν εδώ για την ψηφοφορία. Έκανα λάθος και μπήκα σε λάθος τρένο. Βρέθηκα αλλού. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει έφτασα τουλάχιστον στη συζήτηση και ελπίζω ότι ο συμβολισμός αυτού του λάθους που έκανα, να πάρω λάθος τρένο, να μην είναι καθοριστικός. Εν πάση περιπτώσει, εργάζομαι για τα θέματα αυτά και σε πολλούς άλλους ε, φακέλους και σε άλλες εκθέσεις. Το θέμα του συντονισμού των ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλιξης, παραδείγματος χάρη και των συνεπειών εν ώψη του Brexit είναι κάτι που με έχει απασχολήσει. Δεν άκουσα τι είπε η Ντανούτα, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα θα μίλησε για τους εργαζόμενους ε, που βρίσκονται στην ε, Μεγάλη Βρετανία, όχι μόνο η Πολωνία, ένας μεγάλος αριθμός εξάλλου Πολωνών είναι αποσπασμένοι και το θέμα της επιστροφής τους Ξέρουμε ότι θα προκύψουν πολύ σοβαρά θέματα όσον αφορά τον συνυπολογισμό των δικαιωμάτων μετά την επιστροφή αυτών των ανθρώπων. Βάσει ποιων κανόνων μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης, οι Βρετανοί εργαζόμενοι στην Ευρώπη. Και όχι μόνο οι Βρετανοί, αλλά και αυτοί οι οποίοι από την Βόρεια Ιρλανδία βρίσκονται σήμερα σε ευρωπαϊκές χώρες και εργάζονται στις δικές μας χώρες. Σε περίπτωση λοιπόν σκληρού Brexit, τι ακριβώς προβλέπετε όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων τους και στην περίπτωση της μεταφοράς στην ε, χώρα από την οποία προέρχονται, γιατί δεν πρόκειται όλοι οι εργαζόμενοι σε μια χώρα να ζητήσουν και να πάρουν την ε, υπηκότητα της χώρας αυτής. Επίσης όλα τα ειδικά θέματα που προκύπτουν σε σχέση με την Ιρλανδία. Συγκεκριμένα την Βόρεια Ιρλανδία. Θα πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα ποια είναι η πραγματική θέση που έχει υιοθετήσει η Βρετανική κυβέρνηση όσον αφορά την εκτίμηση των Βρετανών για τις προτάσεις του Μισελ Μπαρνιέ όσον αφορά θέματα που αφορούν την Βόρεια Ιρλανδία, ο συντανισμός των ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για τους ε, κατοίκους της Βόρειας Ιρλανδίας. Αυτό το θέμα σίγουρα είναι εξαιρετικά σημαντικό, πρέπει να το επεξεργαστούμε. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια θέση αρχής Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον εισηγητή και πιστεύω ότι αν δείξουμε ενότητα, αυτό θα είναι κάτι πολύ θετικό. Ευχαριστώ. Ο κύριο Πυρίνσκι θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, mm. Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να επιβεβαιώσω ότι μας ενδιαφέρει να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις από μέρους της Επιτροπής στις ερωτήσεις που έχουν θέσει οι εισηγητές και οι συνεισηγητές. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για τους ε, Βούλγαρους οι οποίοι ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και για τους Βρετανούς αυτούς οι οποίοι έχουν επιλέξει να ζήσουν ε, στη Βουλγαρία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σαφείς απαντήσεις από μέρους της Επιτροπής. Ελπίζω ότι ο κύριος Κοράλε ή οι συναδελφοί του θα μας απαντήσουν. Αν κανείς άλλος δεν θέλει να πάρει το λόγο, μπορώ να δώσω το λόγο στο Γενικό Διευθυντή Κοράλια. Είμαι σίγουρος ότι θα μας ενημερώσει για όλα αυτά τα σημεία τα οποία έχουν θίξει οι διαφορετικοί ομιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνατε για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο βεβαίως εξετάζουμε σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή και το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν πει και έχουν επαναλάβει ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συμφωνήσουμε όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και να λάβουμε υπόψη μας ότι σε μια τέτοια περίπτωση όλα αυτά τα έκτακτα μέτρα δεν θα ήταν ε, απαραίτητα. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να το προϋποθέσουμε αυτό, γι' αυτό και αυτά τα έκτακτα μέτρα είναι απαραίτητα. Είναι επίσης και μονομερή. Αυτή η μονομέρεια αυτών των προτάσεων, αν θέλετε, είναι προφανής και περιοριστική, κυρίως στον τομέα συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί το λέω αυτό. Για να υπάρξει συνεργασία στον τομέα αυτό, χρειάζεται και οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει μονομέρεια, δεν υπάρχει δυνατότητα να μετριαστούν οι επιπτώσεις ε, μιας τέτοιας ε, πράξης. Και καταλαβαίνω πολύ καλά αυτά που είπε η κυρία Λάμπερτ, η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά πολύ καλύτερα από μένα το θέμα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αυτή η εξίσωση είναι πολύ δύσκολο να επιληθεί για όλους αυτούς τους λόγους. Άρθρο 48 εξορισμού. Το άρθρο 48 δεν μπορεί να καλύψει θέματα που αφορούν αρμοδιότητες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία τρίτη χώρα. Από τις 29 Μαρτίου, τα μεσάνυχτα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει μία τρίτη χώρα. Επίσης, το άρθρο 48 δεν μπορεί να καλύψει τα θέματα αυτά που έθεσε η συγγήτρια, η κυρία Χάρκιν, μέσω του κυρίου Καλβέ, για θέματα διαμαχών, συγκρούσεων και πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας. Το 800, ο κανονισμός 843 και οι αρχές της ίσης μεταχείρισης μεταξύ λέει, των Βρετανών πολιτών και των υπολείπων πολιτών της Ευρώπης. Αυτό θα διασφαλιστεί. Δεύτερον, η αρχή της του συνυπολογισμού των δικαιωμάτων όσον αφορά τουλάχιστον την νομοθεσία που εδώ θα πρέπει να εφαρμοστεί για θέματα περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης. Η κυρία Αρκίν αναφέρει επίσης το πεδίο εφαρμογή για το κανονισμό 843. Όχι, δεν μπορεί να επεκταθεί. Έχουμε συμφωνία και αυτό έγινε στην περίπτωση της Τουρκίας. Εδώ όμως δεν υπάρχει συμφωνία, εκτός αν υπογραφεί κάποια συμφωνία. Επίσης η νομική βάση 352 που επιτρέπει την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και για θέματα έκτακτων μέτρων και πολύ περιορισμένης εφαρμογής. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Περιμένουμε κάποια αντίδραση από μέρους των Βρετανών αλλά ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να λάβουν μονομερή νομοθετικά μέτρα και είμαστε σε επαφή με όλους αυτούς. Ο μηχανισμός συντονισμού τώρα. Ο κύριος Μπάλας επίσης γίνεται σιγά σιγά ειδικό για θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Εμείς συνομιλούμε με τους 27, με τα 27 κρατημέλη για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε βάσει όλων αυτών των περιορισμών και να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την κατάσταση. Είδα ότι υπήρχαν και δύο ή τρία άλλα θέματα που έθιξε η κυρία Λαμπέρ, παραδείγματο χάρη. Τι γίνεται με τις ε, θεραπείες οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Εδώ θα εφαρμοστεί το κοινωνικό δίκαιο. Από τα μεσάνυχτα της 29ης Μαρτίου και θεωρούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει θα μπορέσει να συνεχίσει να καλύπτει τα έξοδα αυτά, αλλά δεν υπάρχει νομική υποχρέωση. Ελπίζω, όπως είπε και η κυρία Λάμπερτ, ότι οι πολίτες, ε, οι Βρετανοί πολίτες αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν ε, αποκτήσει και συσσωρεύσει δικαιώματα θα μπορέσουν να τα μεταφέρουν ε, τη στιγμή που θα αποχωρήσουν. Πιστεύω ότι αυτή η νομοθετική πρόταση δεν καλύπτει παρά μόνο ό,τι έχει συμβεί πριν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για οτιδήποτε συμβεί μετά. Όλοι αυτοί οι οποίοι μετακόμισαν πριν την αποχώρηση του, του Ηνωμένου Βασιλείου και είχαν κάποια δικαιώματα βάσει αυτής της, αυτού του καθεστώτος. Ολοκληρώνω και θέλω να σας πω ότι η πρόθεση του Συμβουλίου είναι να ακολουθήσει την διαδικασία του άρθρου 50. Η ειδική ομάδα εργασίας για το άρθρο 50 συνεχίζει τις εργασίες της. Το θέμα είναι κατεπήγον, η διαδικασία είναι επίγουσα και πραγματικά δεν μιλάω εδώ εξ ονόματος του Συμβουλίου και αν ε, υπάρχουν άλλες πληροφορίες ε, μπορείτε να με ενημερώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω απαντήσεις. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω τα μέλη της Επιτροπής μας. Υπάρχουν ε, ερωτήσεις είτε από τους ε, συνεισηγήτρες. Αν όχι, ε, θα ήθελα... Να σας διαβάσω τις αποφάσεις των συντονιστών. Οι συντονιστές καλούν τους συγγέτριες να ακολουθήσουν ε, και να υποβάλουν συστάσεις από τις διαδικασίες. Θεωρούν ότι η τυπική διαδικασία υπό το άρθρο 49 θα ήταν η πλέον κατάλληλη να ακολουθηθεί. Αυτά. Για τον προσανατολισμό που αποφάσισαν να ακολουθηθεί ε, οι συντονιστές. Ε, α, η συνάδελφος Λάμπερτ θέλει το λόγο, παρακαλώ. Ένα σχόλιο που έκανε ένας από τους συναδέλφους γιατί επιλέξαμε αυτήν τη διαδικασία. Επειδή αυτά τα δείγματα, αυτές τις ειδήσει είχαμε από το Συμβούλιο. Ε, όσα περάσαν από το άρθρο 50 δεν είχαν τροπολογίες από το Συμβούλιο, τα του Εράσμους. Οπότε σκεφτήκαμε ότι θα και κατά αυτόν τον τρόπο. Είχαμε τέτοια δείγματα. Äh, Υπάρχει κάποιο παρόν από το Συμβούλιο εδώ που θα ήθελα να τοποθετηθεί από τη Ρουμανική Προεδρία ενδεχομένω. Ευχαριστώ. Δεν έχω εντολή να παρέμβω για την διαδικασία, όμως μπορώ να σας πω ότι είμαι επικεφαλής ε, του τμήματος ΕΠΣΚΟ στην Ρουμανική ε, Αντιπροσωπεία και προεδρεύω αυτό το εξάμεινο στις ομάδες εργασίας κοινωνικών δικαιωμάτων. Δεν θέλουμε ε, παράταση της εντολής ή του κειμένου. Για μας είναι σαφές ότι θα πρέπει να ακολουθεί ταχεία διαδικασία. Και έτσι πρέπει να μείνουν τα πράγματα. Ωστόσο, είναι σαφές ότι στην, στην ομάδα εργασίας του άρθρου 50 ε, θα συζητηθούν τα θέματα αυτά την επόμενη εβδομάδα, οπότε ε, θεωρώ ότι οι προθεσμίες που έχουμε συζητήσει με τις συνεισηγήτριες ανεπίσημα είναι φυκτές και νομίζω ότι θα ακολουθήσουμε ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Οι τροπολογίες ε, θα δυσχεράνουν σημαντικά και ουσιοδός την, την όλη διαδικασία. Äh, Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να ρωτήσει κάτι, όχι. Α, Γκυγιόμ, παρακαλώ. Euh, ναι. Για να είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα αυτά που είπαμε. Η διασύνη του Συμβουλίου επί του θέματος Ε, θα πρέπει να μας οδηγήσει και στο να μην βρεθούμε εξαπρόπτους. Θέλουμε αποτελεσματικές λύσεις για τους πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι σαφώς ε, η, η μόνος τρόπος να εκπροσωπηθούν νομίμως είμαστε εμείς στο Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πλήρη εμπλοκή και ανάμειξη στην όλη διαδικασία για την εξέταση του θέματος, διότι μετά σίγουρα θα υπάρχουν παρανοήσεις που θα μας αποδυναμώσουν εμάς τους ίδιους. Υπάρχει, Τζιν ε, Λάμπερτ, κάποια ερώτηση από την πλευρά σου, έχω καταλάβει σωστά. Μιλάμε για την ομάδα εργασία του άρθρου 50. Δεν είναι το ίδιο με τη διαδικασία 50 βάσει του άρθρου 50 στο Κοινοβούλιο. Να είμαστε τελείω ε, σαφεί ω προ αυτό συμφωνούμε όλοι. Θέλουμε να ολοκληρωθεί όσο πιο γρήγορα και όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα γίνεται. Διότι είναι προς όφελος των πολιτών κάτι τέτοιο. Προς στιγμήν ε, εργαζόμαστε βάσει του 49. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο και μετά θα δούμε τι θα προκύψει και από το Συμβούλιο στι συζητήσει του την επόμενη εβδομάδα. Η πρόθεσή μα σε κάθε περίπτωση είναι να το ολοκληρώσουμε ώστε οι πολίτες να έχουν κάτι να τους καθησυχάζει ως προς κάτι, ακόμη και αν προκύψει το χειρότερο σενάριο και δεν υπάρξει καμία συμφωνία. No deal στις 29 Μαρτίου. Λοιπόν, για την ε, Για τα διαδικαστικά και τις προθεσμίες θα ενημερωθείτε λεπτομερώς με βάση τα όσα θα αποφασίσουν και οι συντονιστές, αλλά νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία ότι θα ακολουθήσουμε την ταχεία διαδικασία ώστε να φωτίσουμε το θέμα αυτό για τους πολίτες μας το συντομότερο δυνατό. Νομίζω ότι υπάρχει ε, συναντήληψη μεταξύ των μελών των, της ε, Επιτροπής μας και των συντονιστών και νομίζω ότι αυτό είναι και ό,τι καλύτερο για τους Ευρωπαίους πολίτες εν ώψη του Brexit. Λοιπόν, να κλείσουμε το θέμα αυτό. Ήταν το τελευταίο σημείο της ημέρης σας διάταξης. Επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 18 και 19 Φεβρουαρίου εδώ στις Βρυξέλλες και σας ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς, ευχαριστούμε και εμείς για την δουλειά τους. Γεια σας.